Μπροκ το έκανε ήδη. Εμένα τουλάχιστον μου είπε ότι ήδη με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου ήρθε σε επαφή και συζήτησε το θέμα αυτής της περίπτωσης. Τώρα, οι αρμόδιες κυπριακές αρχές με ενημέρωσαν για τον διορισμό του συναδέλφου Ιωάννη Κασουλίδη ως Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου από την 1η ε, Μαρτίου. Εξ ονόματος του Σώματος θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Κασουλίδη για τον διορισμό του ως Υπουργό Εξωτερικών της ε, Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύριος Ανδρέας Πιτσιλίδης θα τον αντικαταστήσει από την 4η Μαρτίου. Συγχαίρω τον συνάδελφο Κασουλίδη όπως είπα και καλωσορίζω τον συνάδελφο Πιτσιλίδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7 <clears throat> για την πράξη όσον αφορά τις, ε, την εκλογή μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με το εδάφιο 4, το, το άρθρο 4 ε, από την 1η ε, Μαρτίου 2013 διαπιστώνει την χειρία και της έδρασε και λαμβάνει υπόψη τον διορισμό του συναδέφου Ανδρέα Πιτσιλίδη στην έδρα αυτή από την 4η Μαρτίου 2013. Ο συνάδελφος σύμφωνα με το άρθρο 3 εδάφιο 2 του κανονισμού θα μπορεί να συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στις συνεδριάσεις ε, του Ευρωκοινοβουλίου εφόσον δεν θα έχει ευρεθεί κάποια, ε, κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την εντολή του και εφόσον θα έχει δηλώσει γραπτός ότι δεν έχει κάποιο αξίωμα ή ιδιότητα που να συγκρούεται με την ιδιότητά του ε, ως Ευρωβουλευτού και να καθιστά σύμβατη αυτή την ιδιότητα. Στις 20 Φεβρουαρίου το